εφόσον δεν έχει υπάρξει κάποια ένσταση και υπό την προϋπόθεση ότι η κυρία Σάξα έχει δηλώσει ότι δεν έχει κάποιο αξίωμα το οποίο να συγκρούεται με το αξίωμα της Ευρωβουλευτού και να είναι σύμβατο με αυτό. Η κυρία Αγγέλικα Βέτμαν εγκαταλείπει την κοινοβουλευτική ομάδα της ΑΛΔΕ και από την 8η Απριλίου 2014 θα ανήκει στους μη εγγεγραμμένους. Από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχω κάποια αιτήματα για διορισμού σε αντιπροσωπείες και